η έκθεση Γκούτελαντ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης. Η συγγήτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους χιώδης εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Εδώ έχουμε την απάντηση του Κοινοβουλίου στον πίνακα αποτελεσμάτων για το 2017, το scoreboard ε, που συντάσσεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δίνει την εικόνα της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας των συστημάτων δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2017 προσθέθηκαν και κάποιες νέες πτυχές, παραδείγματος χάρη το πώς έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές ε, σε ε, ε, αποτελεσματικά, σε αποτελεσματικές προσφυγές και νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα μπορούν σιγά σιγά να αποκτήσουν και μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεσή μας εξετάζουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και το πώς αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας το να διασφαλίσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Χρειαζόμαστε ένα δικαστικό σύστημα ανεξάρτητο από πολιτικές επιρροές, ανεξάρτητο από οικονομικές επιρροές και τονίζουμε τη σημασία του ανεξάρτητου εισαγγελέα. Ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να ενισχύσει τη θέση του εισαγγελέα. Καταγράφουμε την έλλειψη δεδομένων σε ορισμένους τομείς και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση ούτω ώστε να έχουμε συγκρίσιμα δεδομένα. Επίσης, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάσει καλύτερα κριτήρια για το πώς τα κράτη-μέλη τηρούν τις αρχές του κράτους δικαίου. Εξετάζουμε παραδείγματος χάρη τα κριτήρια της Επιτροπής και τα συγκρίνουμε με τα κριτήρια των κρατών μελών. Εξετάσαμε επίσης την πρόσβαση των πολιτών στο δικαστικό σύστημα και θα πρέπει ε, να ε, ε, ενισχύσουμε την πρόσβαση και οι πιο ευάλωτες ομάδες να διευκολυνθούν για να έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα. Επίσης ε, καταγράφουμε το ότι το ποσοστό των γυναικών δικαστών έχει μειωθεί σε πολλά κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο στυλιτεύουμε και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την ισότητα των φύλων και στο δικαστικό σύστημα. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Προτείνουμε τη βελτίωση της εκπαίδευσης των δικαστών και να δίδεται ειδική κατάρτιση για τα στερεότυπα που έχουν σχέση με τα φύλλα. Θα χρειαστεί ένα πίνακα αποτελεσμάτων ευρύτερο που να συμπεριλαμβάνει και κάποιε δικαστικέ ε, διαδικασίε και προτείνουμε ένα νέο δίκτυ να προσθεθεί η πρόσβαση ε, το δικαστικό σύστημα ατόμων εναντί των οποίων ε, υφίσταται διακριτική μεταχείριση διότι ανήκουν σε συγκεκριμένε ομάδε. Σημαντικό ρόλο επίσης ε, για την προστασία των καταναλωτών θα παίξει και το να ληφθούν υπόψη οι συλλογικές προσφυγές. και να του δίνεται η δυνατότητα, στους καταναλωτές, να δίνεται η δυνατότητα ε, αποζημίωσης. Εναλλακτικοί ε, μηχανισμοί ε, επίλυσης διαφορών. Και αυτά μπορεί να περιληφθούν στον πίνακα αποτελεσμάτων των συστημάτων δικαιοσύνης κατά την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική συνεργασία και ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα συμπεράσματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο στα πλαίσια του ΚΑΤΣΤΙΑΙ ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη είναι οπωσδήποτε θεμελιώδου σημασίας. Όμως ιδίως στην Ελλάδα βάλεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρύθμιση στο μνημόνιο που λέει ότι εάν εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει τα δημοσιονομικά μέτρα που επιβάλλονται από το μνημόνιο τότε οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος. δηλαδή η ίδια η τρόικα επιβάλλει με τον τρόπο αυτό μέσω των μνημονίων την μη τήρηση των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης. δεύτερον η πρόσφατη παρέτηση του προέδρου του συμβουλίου της επικρατείας στην ελλάδα αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη ότι πλέον κλονίζεται ο θεσμός της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στην ελλάδα. οφείλει η έκθεση να εξετάσει το πώς λειτουργεί η τρόικα και το πώς επί της ουσίας διαλύει κάθε έννοια ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη που βρίσκονται κάτω από την τρόικα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάτολα, η αντιπρόεδρος Χάτολα έχει το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Χάτολα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κούτελάντα, την εισηγήτρια, για την έκθεσή της και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ζητάει από την Επιτροπή η έκθεση στη συγκριτική, στο συγκριτικό εισχύρημα να χρησιμοποιήσει και να συμπεριλάβει και τις συλλογικέ προσφυγές, γιατί είναι κάτι πολύ βασικό και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό και έχει δημοσιοποιήσει νομοθετική πρόταση από αυτού όσο εμείς δουλεύαμε πάνω σε αυτή την έκθεση. Η νομοθετική πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συλλογικέ ε, προσφυγές όμως τι κάνει. Λέει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέσω επίλυσης και θα καταργούσε ε, φραγμούς για πρόσβαση στην δικαιοσύνη το σύστημα αυτό των συλλογικών προσφυγών. Θα πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό για επιχειρήσεις ή οργανώσεις που έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, συχνά εξαιτίας κάποιων τεχνικών ζητημάτων ο κόσμος τελικά δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη καθόλου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαδρίδης έχει το λόγο. Ε, θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για την έκθεσή τους, όμως θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ομοιογένεια στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των κατευθυντήριων γραμμών από το ευρωπαϊκό δικαστήριο και αναφέρομαι ειδικότερα γιατί έχω προσωπική αντίληψη των αποφάσεων που αφορούν τον τραπεζικό τομέα και είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να επανεξετάσουμε διότι η ανομοιογένεια στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων πλήττει και την έννοια της απονομής της δικαιοσύνης αλλά πλήττει και πολλά άλλα θέματα όπως είναι για παράδειγμα ο αθέμητος ανταγωνισμός. το δεύτερο σημείο και τελειώνω είναι ότι θεωρώ πως έπρεπε να υπάρχει έστω και μία πρόταση που να καταγράφει στην έκθεση ότι στο βόρειο κατεχόμενο μέρος της κύπρου που είναι μέρος της ευρωπαϊκής ένωσης δυστυχώς δεν εφαρμόζεται το κράτος δικαίου διότι το εμποδίζει ο τουρκικός στρατός. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα το λόγο έχει η Επίτροπος Μπούλκ. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Ευχαριστώ ε, την εισηγήτρια, κυρία Γκουδελέ και το Κοινοβούλιο για την ε, ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Είναι θεμελιώδου σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, για την κοινωνική ειρήνη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε από την Επιτροπή, ο πίνακα αποτελεσμάτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το προηγούμενο έτος ε, και χαίρομαι που λαμβάνεται υπόψη πολλά από τα στοιχεία. Ο πίνακα αποτελεσμάτων είναι ένα εργαλείο το οποίο βελτιώνεται συνεχώς και οι συστάσεις σα θα ληφθούν υπόψη για το μέλλον. Η έκθεσή σας ζητεί την επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, με τον πίνακα αποτελεσμάτων και στην ποινική δικαιοσύνη. Το 2016 επεκταθήκαμε και στο ξέπλυμα χρήματος και ε, για όλες τις χώρες αναγράφονται οι ε, υποθέσεις ξέπλυμα χρήματος. Η πρωτόδικη διαδικασία παίρνει περίπου ένα χρόνο κατά μέσο όρο και σε ορισμένα κράτη-μέλη μέχρι δύο χρόνια. Ζητάτε επίσης ε, να ενισχύσουμε την αυτονομία ε, του Ευρωπαίου Σαγγελέα. Ε, ο πίνακα αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι για πρώτη φορά δείχνει τώρα πώς είναι οργανωμένες οι εισαγγελίες στα κράτη-μέλη. Ο πίνακα αποτελεσμάτων ενισχύει τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξαμήνων. Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εθνικών πλαισίων και των ε, νομικών δικλείδων σε στενή συνεργασία με τα δίκτυα των δικαστών. Και έχουμε μια μέτρηση της ανεξαρτησίας ε, της δικαιοσύνης όπως εκτιμάται από τις επιχειρήσεις και από το κοινό. Τονίζουμε τη σημασία των εργαλείων τεχνολογίας πληροφορικής στις δικαστικές διαδικασίες και την δυνατότητα πρόσβασης σε δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά. θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα ε, και σε άτομα με ειδικές ανάγκες ε, όπως ε, άτομα με τυφλούς ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα θα ληφθούν υπόψη και οι δημόσιε διαβουλεύσει για τα, τον επόμενο πίνακα αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι ε, μία από τις βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορική είναι η συγκέντρωση δεδομένων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο που ζητά από τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν εξετάζουμε οποιοδήποτε νέο τομέα θέλουμε να καλύψουμε, θα λάβουμε υπόψη τους στόχους που έχει ο πίνακας αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα κράτη-μέλη με βάση ένα ξεκάθαρο δίκτυο, ο οποίο θα είναι προσαρμοσμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, το ψήφισμά σα φτάνει σε μια χρονική στιγμή που ε, είναι υψηλή προτεραιότητα ε, στο θεματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα που συζητάμε και τα θέματα τη δικαιοσύνη. Θα συνεχίσει ο πίνακα αποτελεσμάτων να εξελίσσεται για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ανεξαρτησία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού του συστήματο, πράγμα το οποίο είναι κέρια σημασία για την τηρήση του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπε, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε, αύριο θα γίνει η ψηφοφορία.